I think we can start. Ja, schönen guten Morgen. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίες μου και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών ε, που έχει καλέσει ο κύριος Κοχ ε, από ε, την πόλη του, την Ερφούρτη, εκπρόσωποι των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων της Bundeswehr. Καλωσορίσατε θερμά στην Επιτροπή μας. Ερχόμαστε λοιπόν αμέσως στις ψηφοφορίες στην έκθεση Ζάκη Φώστερ για τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να κάνουμε ένα τεστ πρώτα, να δούμε τα μηχανήματα δουλεύουν. Άρχεται η ψηφοφορία. Να μην την κλείσω ακόμα. Ε. Το σύστημα λέει ότι είναι εντάξει. Μπράβο, συγχαρητήρια Βιμ Βαντεκάμπ. Ο Γιάννης Νίλσον έχει ξεχάσει την κάρτα του, αλλά το λαμβάνουμε υπόψη. Στα ρουμανικά υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία, κάποιο τεχνικό μάλλον. Να το δοκιμάσουμε και πάλι. Μπορείτε να μας πείτε αν είναι εντάξει, ακούτε τίποτα ρουμανικά. Όχι. Σε στήνα σας. No? Er sagte, er hätte keine. Also in dem Raum haben wir keine 22 Sprachen, sondern nur 16 oder so. Aha. war das denn angekündigt? Uh, We have only 16 languages. 16 γλώσσες έχουμε μόνο και σήμερα δεν υπάρχουν ρουμανικά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν εξαρτάται από τη θέλησή μας, εξαρτάται από την αίθουσα. Μόνο 16 καμπίνε διερμηνία έχει αίθουσα. Το καταλαβαίνω και δέχομαι την εξήγησή σου, αλλά είμαστε δύο τακτικά μέλη στην Επιτροπή από τη Ρουμανία και είναι φυσιολογικό να έχουμε ε, τη γλώσσα μας. Και είναι η μόνη επιτροπή στην οποία δεν έχουμε ε, διερμηνία στα ρουμανικά. Ωραία, θα το ελέξουμε και σήμερα κάτι εξαίρεση, δεν είναι για πάντα αυτό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 40 υπε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 46 Πέρασε. απορρίπτεται 25 κατά 16 υπέρ 47 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Από τη Λίμπη 4 στη παράγραφο 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ για την ε, τροπολογία παριθμών 63. Άρχεται ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. Πέρας. Abgelehnt. Amendment. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 της Λίμπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η έντεκα της ε, ελευθερίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 73. Ε, α, έχει ε, αποσυρθεί 74 υπέρ Split vote υπέρ της 74, πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίφθεται. Τσεκ, πολύ ωραία. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν τσεκάρουμε της τροπολογίας 74. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 21-21 ισοψηφία. Αλλά έχουμε και άλλη μία ψήφο κατά χωρίς κάρτα. Απορρίπτεται λοιπόν. Άρα πολύ προσεκτικά το είδα. Η συμβιβαστική 6 είπε, Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 82 υπέρ. εκεί Κατά αποχές το ελέγχουμε 82 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τοπολογία κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 87 υπέ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική παριθμόν 7 εδώ υπάρχει ένα λάθος γιατί η Γκουε δεν συμφωνεί με το συμβιβασμό αυτό. είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 94 ψήφι πέ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 8 είπε. κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο ε, ναι, λέει ο Πρόεδρος, έχουμε μια προφορική τροπολογία. Ε, Ένα είναι κατά, δεν φτάνει. Τρει τρεις πρέπει να... Ε, ναι, σηκωθείτε όμω. Πρέπει να εγερθείτε, λέει, για να σα δουν όλοι. Ωραία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την προφορική τροπολογία, άρα ψηφίζουμε χωρί την προφορική ψηφιπέ. Α, όχι, έχει καλυφθεί λοιπόν από το συμβιβασμό, δεν χρειάζεται άλλη ψηφοφορία. Πάμε στη ΛΥΜΠΕ 9, υπέ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Παράγραφος 20, προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την 20 παράγραφο με την τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές αυτό θέλει έλεγχο. Στην 127 παρακαλώ, άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 31-11 εγκρίνεται και άλλοι δύο. άλλο άλλος ένας, 31-11, συγγνώμη. 128 υπέρ. Κατά. Ναι, ναι. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 130. Όχι. 132 τότε. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 133. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται 141 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 143 υπέρ Καταπίπτει. 142 επίσης. Τότε πάμε στην 145. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ τι θέλετε, έλεγχο για την 7 τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρασε. Ισοψηφία 22-22, 23 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 151 παρακαλώ αρχίζει τώρα η παλήθευση. Πέρας. 19 υπέρ. 20 υπέρ. 25 κατά. Απορρίπτεται. Λίμπε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίπε 12, θέλετε έλεγχο. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 23 δηλαδή υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 13 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 13 της Λίμπε αρχίζει ο έλεγχος. Ist geschlossen. Πέρας. 17, 18 υπέρ, 27 κατά απορρίπτεται. Λίμπε 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 153 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11. Έχουμε εδώ προφορική της κυρίας Γοβονταλών. Ε, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θέλω να αλλάξουμε το τέλος τροπολογίας αυτή να μην βούμε ένα χωριστό ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά διαφορετικές διατάξεις στο ίδιο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Διαφωνεί κανείς? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε την 11 με αυτή την προφορική τροποποίηση. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. 24 υπέρ 20 κατά εγκρίνεται. Μάλιστα. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, ας το ελέγξουμε λοιπόν. Γιατί 12 αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρα. 20-22 23 δηλαδή. 13. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 25. Ψηφιπέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26 Υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 Υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 Υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 Υπέ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία παριθμών 1 ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία είναι και ονομαστική. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 44. 45 υπέρ. Ένας κατά. Καμία αποχή εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια Τζάκη Φώστερ. Okay, Όπως βλέπω, υπάρχουν ελεύθερες θέσεις. Γι' αυτό στέκονται όμως ορισμένοι επισκέπτες. Μήπως να καθίσετε παρακαλώ για να μπορέσετε να ακούσετε και τη διερμηνία. Αν έρθει βέβαια κάποιο συνάδελφο, έχετε προτεραιότητα στι θέσει των ε, απόντων. Μπορείτε να καθίσετε για να ακούτε και τη διερμηνία. Εδώ βλέπετε πόσο χώρο έχει. So, wir kommen jetzt zu der nächsten Abstimmung. Λοιπόν, επόμενη ψηφοφορία, νέε προκλήσεις και έννοιες για την πρόθεση του τουρισμού στην Ευρώπη. Η συγκήτρια είναι η κυρία Ζαμπέλα Ντεμόντε και προχωρούμε στην ψηφοφορία. Η πρώτη είναι μια προφορική τροπολογία, διαφωνεί κανείς. Α, όχι, αμπλόκ λέει εδώ, Όλε τι συμβαστικέ. Όλε οι συμβαστικέ ψηφίζονται μαζί, 1, 3, 4, 5, 6 και 13 όχι έξτρα. Οι υπόλοιπε είναι unblock. Είναι μεγάλη πρόκληση είπε. αλλά θα κερδίσουμε πολύ χρόνο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το σύνολο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παράγραφος ε, πρώτη, προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανεί. Όχι. Ψηφίζουμε αυτή την προφορική ψηφή Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 50. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική ενα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 24 υπέρ κατά αποχές απόρριψη. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε έλεγχο για την 54, αρχίζει. Παόλ. Πέρας. 17 υπέρ 27, κατά απορρίψετε. Η τροπολογία 55 λοιπόν είπε; Ορίστε. Oh, 55. 55. Κάτι λέει η κυρία Φώστερ εκτός μικροφώνου, δυστυχώς δεν ακούγεται. Okay. Τι θέλετε, να επαναλάβουμε την ηλεκτρονική στην 54 παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρα. 23 υπέρ, 22 κατά εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Η 56 υπέρ. Καταπίπτει, συγγνώμη. Η 57 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 58 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 είπε. Κατά. Αποχέ... Α, την ελέγχουμε. 59. Άρχεται ψηφοφορία. Και λίγη. ναι, υπέρ 33 κατά. Ένα μυστήριο πράγμα. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 11 υπέρ. Καταπέφτει. Α, εντάξει, έχει διεκπαιρωθεί. Προφορική τροπολογία 2. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Όχι. Wer ist dafür? Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 76. 76 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 3 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Η 83 υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 84. Καταπίπτει. Η 111. Υπέρ, ε, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση 107 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. 16 με 28 απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 117 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 120 καταπίπτει, η 119 επίσης, η 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 128 καταπίπτει. Πάμε στην 133 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό παρακαλώ. Next. Ah, λοιπόν, ε, ξεχάσαμε μία τροπολογία, την 129. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και την 131 επίσης, γιατί δεν εγκρίθηκε η 126, η 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα πάμε στην 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 2 υπέρ. Μισό λεπτό. Η κουλτ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κουλτ 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κουλτ 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κουλτ 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κουλτ 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ΙΜΚΟ 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η Κούλτ 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η Κούλτ 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η κουλτ 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η κουλτ 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονική επαλήθευση η 157 ψηφίζουμε παρακαλώ λοιπόν 157 ψηφίζουμε έκλειση ψηφοφορία Απορρίπτεται. Η 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 159 παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφορία. 31 31-13 εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12, προφορική τροπολογία, διαφωνεί κανείς με την προφορική, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 22 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 22 της Επιτροπής Πολιτισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 32-11 εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 32. Ορίστε τι θέλετε. πίπτη. Όχι. 169 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 κατά πίπτη, όπως και η 177 όχι όχι 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΕΜΚΟ 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 18 Α, μια στιγμή έχει καταπέσει μάλλον. Κουλτ 38 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 74. Τι γίνεται με την 74 υπέρ του συνόλου κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 147 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αριστα. Βάλα 215 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίψη 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίψεται. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 249 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούλτ 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 244 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 259 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για τη 259. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24-21 εγκρίνεται. 262 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο καταπίπτει 2,60 επέ. κατά αποχές απορρίπτεται. 2,61 επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 278 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 280 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 283 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 16 είπε κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την Ήμικο 16 αρχίζει τώρα. Πέρας. Τι έγινε, απερίφθη. Ήμκο 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 313. 313 κατά πίπτη. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 315 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 316 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 317 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ίμκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 300 oral amendment ε, 4. Η προφορική τροπολογία 4 στην παράγραφο 29. Διαφωνεί κανεί, όχι. ψηφίπε Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 325 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 327 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ήμκο 9. πίπτη. 331. Ψήφι Π. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 232 επέ. Κατά. κατά, Απορρίπτεται. 334 ΥΠΕ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 340 ΥΠΕ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 29 ΥΠΕ. Κατά. απόχε. Εγκρίνεται. 349 υπέρ. Κατά. άποχε, Έλεγχος. Για την 349. Άρχεται η ψηφοφορια περα Πέρας. 22-22 ισοψηφία. Απορρίπτεται. 3.35 υπέρ κατά άποχες δεν ψηφίζεται 335 παρακαλώ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 3.37 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 350 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε σε αιτιολογικές σκέψεις, recitals. Όχι, είναι συμβαστικά, τα έχουμε ψηφίσει αυτά. Α, πάμε στην 6. Α, τον κύριο Ρικέ ξεχνάμε, είναι δυνατόν. 6 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, το άλλο... 23 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. 24 είπε, και τα υπόλοιπα μαζί είπε μέχρι και την 27. Κατά αποχή εγκρίνεται. 27 όχι. Α, τώρα 27 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ. Κατά. Φαίνεται σαν να έχει απορριφθεί, αλλά χρειάζεται έλεγχο. Ε, ψηφίζουμε την 30. Πέρα. 20-24 απορρίφθηκε. 36 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Όχι, καταπίπτει. Η 46 λοιπόν. ψηφιπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 ειπε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 ειπε Κατά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 Συγχαρητήρια θερμά κυρία Δεμόντε μου. Ευχαριστώ. <laughs>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 Ich glaube, wir können jetzt weitermachen. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ε, καθίστε και συνεχίζουμε.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 12 κατά κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και ανάγκη για μία στο 9 μάλλον, στο 9 η κυρία Κίλενεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συχνά δεν συμφωνώ με τον Jean-Claude Juncker για πολλά θέματα, αλλά να θυμηθούμε αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο όταν μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Είπε κάτι το οποίο μπορώ να αποδεχθώ, ε, ζήτησε μια Ευρώπη πιο ανθρώπινη και πιο ανοιχτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω μια Ευρώπη που δεν θα βοηθά όσους χρειάζονται. Αν αφήσουμε τους αρχηγούς κρατών να κάνουν τις εθνικιστικές τους πολιτικές, τι θα μείνει από την Ευρώπη. Τίποτα. Οι πρόσφυγες έρχονται από ζώνες κρίσεων, συγκρούσεων ε, της Αφρικής ε, και είναι ένα θέμα διαφιλονικούμενο για την εξωτερική μας πολιτική. Χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις ε, σε περιπτώσεις σημαντικών κρίσεων. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε και να αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει. Όταν υπάρχει μια κρίση πρέπει γρήγορα να αποφασίζουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των μεταναστευτικών ροών που είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι περαστικό αλλά θα επιδεινωθεί και θα επιδεινώσει και ε, την κατάσταση της χώρες όπου η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν συγκρούσεις ε, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική ε, καλό είναι να βελτιώσουμε τις, ε, τη ζωή των ανθρώπων επιτόπου, αλλά δεν πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες μας. Σε ένα φορτηγό στην Αυστρία βρήκαμε ε, ε πρόσφυγες που πέθαναν από ασφυξία. σε πολλά τρένα βρίσκουμε πρόσφυγες που πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη κάνουν ε, ό,τι μπορούν σε πολλά ε, σημεία οι αρχές των κρατών μελών για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες αυτούς, ε, όμως όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό εγώ έχω, έχω συντάξει ένα σχέδιο έκθεσης για το θέμα των θαλασσίων μεταφορών και της ασφάλειάς τους. Νομίζω ότι δεν, δεν απουσιάζει η ευαισθησία από την έκθεσή μου. Πρέπει να έχουμε μια συνολική προσέγγιση για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο κύμα αντιδράσεων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ε, δίκτυα ασφαλείας ε, από τους ίδιους τους πολίτες όταν οι αρχές δεν μπορούν να αναλάβουν τις ε, υποχρεώσεις τους οι πολίτες ακόμη ε, έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Δεν μπορούμε να δεχθούμε όμως ότι τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκοί ε, θεσμοί ε, θα αποποιηθούν των ευθυνών τους και θα βασίζονται στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, στις επιχειρήσεις και στον κάθε ιδιώτη. Κάτι πρέπει να γίνει όταν υπάρχουν ναυάγια στην περιοχή της Μεσογείου. και στα επιβατικά πλοία αλλά και στα ε, πλοία μεταφορών αγαθών και εμπορευμάτων, τα εμπορευματικά πλοία, ε, υπάρχουν υπηρεσίες διάσωσης, επιχειρήσεις διάσωσης. Ε, μέχρι το τέλος του μήνα Ιουλίου πάνω από 130 επιχειρήσεις διάσωσης έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Ιταλίας. 15.000 άτομα ε, σώθηκαν από τις, κατά τις επιχειρήσεις αυτές διάσωσης. Ε, τα εμπορικά πλοία πάνω από 15% ε, των ατόμων που σώθηκαν στα ανοιχτά της Ιταλίας ε, τις έσω, τα έσωσαν εκείνα τα εμπορικά πλοία. Πρέπει όμως να κάνουμε πολύ περισσότερο γιατί είναι τεράστια αριθμή. Σας υπενθυμίζω το δίκαιο της θάλασσας αλλά και τη σύμβαση της ε, ε, διάσωσης της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Ο πλοίαρχος ενός πλοίου, ο καπετάνιος, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει ανθρώπους που ε, βρίσκονται στη θάλασσα και που κινδυνεύει η ζωή τους και να συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης ε, ε, στο βαθμό που δεν δημιουργεί αυτό πρόβλημα ούτε θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του πληρώματός του και των επιβατών. Όμως δεν υπάρχει απαραίτητος εξοπλισμός, ούτε τα πληρώματα είναι καταλήλως εκπαιδευμένα για τις επιχειρήσεις αυτές διάσωσης, Εξού και ο κίνδυνος ασφάλειας που τίθεται για τα πλοία αυτά και για το πλήρωμά τους. Συχνά στα πλοία αυτά ε, δεν υπάρχει αρκετό πόσιμο νερό, δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για την υποδοχή πολλών ε, ατόμων, κάτι το οποίο ορισμένες φορές έχει οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Συχνά Πολλές φορές μέχρι και τα εμπορευματικά πλοία έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις ε, διάσωσης. Τα πλοία αυτά δεν έχουν ε, επαρκή εξοπλισμό, ούτε κατάλληλη εκπαίδευση για τα πληρώματά τους, ε, για την αντιμετώπιση ατυχημάτων ή για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ανθρώπων. Υπάρχουν περιπτώσεις εμπορευματικών πλοίων με χημικές ουσίες ε, που ε, αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα υπάρχει περίπτωση οικολογικής καταστροφής. Η κατάσταση έχει ως εξής. Είναι σαν να πηγαίνει κανείς το πρωί στη δουλειά του. Βλέπει κανείς έναν πεζό, ο οποίος έχει υποστεί ένα ατύχημα. Είναι προφανές ότι θα πάτε να τον βοηθήσετε όσο μπορείτε ε, και θα καλέσετε βοήθεια. Αν όμως αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε μέρα όταν πηγαίνετε στη δουλειά σας και όταν καλείτε τις αρχές σας λένε ότι δεν έχουν επαρκή σπόρους για να μπορέσουν να έρθουν και σας ζητούν ε, να μεταφέρετε εσείς τον ε, τραυματία στο ε, νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο είδους σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Η μόνη λύση είναι περισσότεροι πόροι για τις επιχειρήσεις διάσωσης για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα των προσφύγων για την ασφάλεια και των πλοίων πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο ε, πρέπει να ε, αποβιβάζονται ε, στα ε, λιμάνια για να μπορούν να ε, ζητήσουν άσυλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σύστημα παρακολούθησης και πληροφόρησης σε σχέση με τα πλοία που πλέουν στις ευρωπαϊκές ζώνες και επίσης να υπάρχει συνεργασία με την ακτοφυλακή προκειμένου να είναι πιο ασφαλείς οι θαλάσσιες μεταφορές. Τα μέτρα πρέπει να τα απαραίτητα ε, μέτρα πρέπει να ε, εκμεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερες ε, περισσότερα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων διάσωσης. Πρέπει να κινητοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτικές για την εξασφάλιση και της ασφάλειας αλλά και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών. Πρέπει επίσης ως Ενωμένη Ευρώπη να έχουμε ένα κοινό μέτωπο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ε, κάτι το οποίο έχει ε, γίνει πλέον ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, ε, σαν τους λαθρεμπόρους όπλων που κερδίζουν εκατομμύρια από, αυτή, από αυτό το εμπόριο οι άνθρωποι μάλιστα που έχουν ε, την περισσότερη ανάγκη, τη μεγαλύτερη ανάγκη δεν μπορούν καν τελικά να ζητήσουν άσυλο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και τις εργασίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε καλές προτάσεις ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να συνεργαστούμε καλά και επικοδομητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους σκιώδους εισηγητές και τις πολιτικές ομάδες ε, για τις εργασίες ε, που είχαμε μέχρι σήμερα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση. Ο κύριος ε, Πασκάλ έχει το λόγο. Λουίς Δεγκράντες, Πασκάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια πάρα πολύ για την ευγένειά να αναφερθεί στους και τους και να τους καλέσει ε, σε μια προκατακτική φάση. Και λεπτότητα δείχνει αυτό και ευγένεια και πολιτική ευαισθησία και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Ωραία. Μιλάμε για τη Μεσόγειο, έτσι. Μπορεί να σας φαινόταν αυτό ε, μακρινό και αυτό που είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος για τρομερό όνειδος και έσχος αλλά τώρα αυτό έχει φτάσει σε όλη την Ευρώπη αυτό που κάποιοι θεωρούσαν μακρινό και άσχετο με τις χώρες τους τώρα έχουν καταλάβει ότι αφορά όλη την Ευρώπη η κατάσταση και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αποσπασματικά πράγματα που δεν επιτρέπεται κιόλα. Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσει που λαμβάνονται τώρα σε θεσμικό επίπεδο. Όλα αυτά είναι προφανή και αυτονόητα. Οπότε, καλά είναι αυτά που λέμε, αλλά εμείς γνωμοδοτούμε μόνο. Καμιά φορά υποκύπτεις στον πειρασμό να κάνεις γενικότερες τοποθετήσεις για την ελευθερία, για την αλληλεγγύη, για διάφορα συγκινητικά. Αλλά εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και θα πρέπει στο πλαίσιο το δικό μας αρμοδιοτήτων να συνεισφέρουμε για να βοηθήσουμε στις λύσεις, να δούμε τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε από το δικό μας μετερίζει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τη λύση που δίνεται στο γενικότερο πλαίσιο των ελευθεριών μεν. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να ε, συγκρουστούμε με το Frontex, που βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθεί, αλλά θα πρέπει να ε, φτύνουμε μία έκκληση σε ένα οργανισμό που είναι πάρα πολύ ικανός, όπως είναι η ΕΜΣΑ, για την ασφάλεια στη θάλασσα, ε, είδαμε τι έκανε στην καταπολέμηση της ρήπανσης, ας πούμε, με μεγάλη επιτυχία, που είχαμε ε, πλοία ε, stand-by για να μπορέσουν να να βοηθήσουν και αυτά που είπε τα ωραία λόγια η για τα εμπορικά πλοία ότι είναι υποχρεωμένα μα είναι πολύ θετικό αυτό να τρέξουν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ε, θα πρέπει να έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να το κάνουν θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον Οργανισμό λοιπόν για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, να δούμε μήπως πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων ή εντό των αρμοδιοτήτων του να χρησιμοποιηθεί ω εργαλείο για να συνεισφέρει στι αποφάσει για την έρευνα και διάσωση αυτών των κατατρεγμένων, αυτών των, των, των καημένων πραγματικά που είναι πρόσφυγες και τρέχουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από ε, το θάνατο και πεθαίνουν από την πείνα. Ελπίζω αυτή η άρση του Σέγγεν να είναι απολύτως προσωρινή, αλλιώς θα πέσουν τα θεμέλια της Ευρώπης. Καλή λοιπόν η αλληλεγγύη, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε μια στιγμή να καθίσουμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα συμμετέχουμε στη συζήτηση, αλλά πάντα σας λέω από τη σκοπιά των μεταφορών. Εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για τη λύση του προβλήματος. Τέτοιες τροπολογίες θα κάνουμε εμείς. Να δούμε πώς ε, θα προστατεύονται τα εμπορικά πλοία που πρέπει να βοηθούν. Να ζητήσουμε από τον οργανισμό ΕΜΣΑ να κάνει προτάσεις για λύσεις, χωρίς να συγκρουστεί με τη Frontex γιατί είναι πραγματικά τραγική αυτή η έξοδος. Σήμερα είναι στη Μεσόγειο, αλλά κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις όχθες της Μεσογείου. Και κάποιοι που το βλέπανε μακρινό κατάλαβαν όταν ήρθε στην αυλή τους τι σημαίνει αυτό. Τι γίνεται στη σύραγγα, στη μάχη. Σιγά σιγά έχουν το ίδιο πρόβλημα και στην ξηρά αυτό που έχουμε εμείς στη Μεσόγειο. Όταν αρχίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα στη Μεσόγειο μπορεί να ήταν μεμονωμένο και αποσπασματικό σήμερα είναι απολύτως αποφασιστικό. Και το πρόβλημα είναι για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο για τις μεσογειακές χώρες. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και να το εντάξουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο προσφυγικό, μεταναστευτικό που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει. Με αλληλεγγύη αλλά και με λογική. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριο Κύρκο, παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κιλόνεν γιατί και μέχρι μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε αλλά και όπως μας είπε και από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση που θα περιέχει όλα τα σημαντικά στοιχεία πάντα από το πρίσμα της Επιτροπής Μεταφορών. Και εδώ συμφωνώντας με τον κύριο Πασκουάλ ε, θέλω να πω πως όντως η δικιά μας οπτική είναι η προστασία των πλοίων, των πληρωμάτων, των εμπορευμάτων τα οποία διασχίζουν τη Μεσόγειο. Η κυρία Κελώνη μας είπε πάρα πολύ καθαρά το βάρος που σηκώνουν τα εμπορικά πλοία που διατρέχουν τη Μεσόγειο. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Δεν μπορεί δηλαδή τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να φορτώνει στα εμπορικά σκάφη το ρόλο της ε, διάσωσης έρευνας και διάσωσης των προσφύγων. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει και με τη δική μας έκθεση να δουλέψουμε ώστε ιδανικά να μην κάνουν καθόλου διάσωση παρά μόνο σε ακραίες συνθήκες στη Μεσόγειο τα εμπορικά πλοία και η διάσωση εκτελείται από αυτούς που έχουν την υποχρέωση της, δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Ε, Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στο ρόλο των σκαφών. Είπε ο κ. Πασκουάλη για την έμψα που είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε την άποψή τη. Είναι και η οδηγία 2001 του 51 που δεν έχει ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο και καμιά φορά οι κυβερνήτε των σκαφών βρίσκονται αντιμέτωποι με άλλα προβλήματα όταν προβούν σε εθελοντική διάσωση. Η συγγήτρια σωστά ζητάει να αυξηθούν οι άμεσε δράσει, όμω πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μόνιμη δράση και να εξασφαλιστούν όλοι οι πόροι για μια μόνιμη έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο, γιατί το ζήτημα δεν θα τελειώσει, δεν είναι προσωρινό. Το ζήτημα, όπω βλέπουμε, είναι πολύ ευρύτερο και οι απαντήσει τη Ευρώπη πρέπει, μια και περνάει και από εμά μια γνωμοδότηση, να κοιτάνε και προ το μέλλον. Ε, μερικά ακόμα σημεία μπορεί να είναι η συνεργασία με τις χώρες, τις παράλληλες χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μπορούμε να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και να δώσουμε μια διάσταση ότι όσο καλύτερη συνεργασία υπάρχει με αυτά τα α, μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Τουρκία ας πούμε, που δεν είναι failed state όπως είναι η Λιβύη, τόσο θα περιορίζεται το βάρος που πέφτει στην εμπορική ναυτιλία. Πάντα από το δικό μας πρίσμα της Επιτροπής Μεταφορών όπως επίσης και το πρόβλημα της άμεσης στήριξης των κρατών της πρώτης γραμμής που και αυτό οδηγεί σε καλύτερη έρευνα και διάσωση, άρα σε μικρότερο βάρος στα εμπορικά μας σκάφη. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις ε, μας έχουν κάνει να μιλάμε ήδη για πράγματα που είναι μακριά από την πραγματικότητα. Μιλάμε για διάσωση, μιλάμε για έρευνα και διάσωση των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι ήδη έχουν μπει στα σκάφη, των προσφύγων, που θα έχουν ένα ευρωπαϊκό σπίτι, όπως ήταν και η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου και ελπίζουμε και οι επόμενοι ακόμα πιο πολύ σε βάθος, αλλά έχουν ήδη μπει σε σκάφη, ήδη περνούν, τρέχουν τη Μεσόγειο. Η απάντησή μας και η προτροπή πρέπει ακριβώς για να ε, ελαφρύνουμε πάντα από τη μεριά της Επιτροπής Μεταφορών, να ελαφρύνουμε το βάρος έρευνας και διάσωσης του εμπορικού στόλου, πρέπει αυτές οι κινήσεις να γίνουν από εκεί που ξεκινούν οι πρόσφυγες. Αφού έτσι και αλλιώς θα τους υποδεχθούμε στην Ευρώπη, πρέπει οι κινήσεις να μην τους εμπλέξουμε στα δίκτυα των, ε, λαθρομετα... των εμπόρων, αλλά να τους μεταφέρουμε από εκεί που ξεκινάνε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ρόζα Τόμας, έτσι. Thank you. Um... Ευχαριστώ. κροατικά είναι ο λόγος μου, αλλά επειδή δεν υπάρχουν κροατικά, θα προσπαθήσω πάρα πολύ να κάνω τα σχόλιά μου στα αγγλικά. Ο αριθμός των μεταναστών που περνούν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρώπη είναι πάνω από 300.000 άτομα, τουλάχιστον αυτή τη χρονιά. Ε, και 2.000 214.000 άτομα το 2014. Βλέπετε τα ε, τεράστια αυτά νούμερα που είναι ανησυχητικά και ε, που πρέπει να ε, μας καταστήσουν πιο προσεκτικούς, να είμαστε και πιο προληπτικοί στην αντιμετώπιση μας για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μακροχρόνιες ε, λύσεις ε, αντί για ε, συγκυριακές λύσεις επιτόπου. Πρέπει να ε, δούμε πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ε, προσπαθώντας ε, να διασχίσουν τη Μεσόγειο και πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει στα πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια. Πρέπει επίσης να εντείνουμε τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Ζήτω συγγνώμη, λέει ο... Ζητώ συγγνώμη, λέει Μιλήτρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφράζω έτσι από τα κροατικά ε, στα αγγλικά. Ε, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που κάνουμε ως τώρα. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο όλων των σκαφών, να αυξήσουμε την, ε, τον έλεγχο ασφαλείας και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δικαιότερη προς όλες τις πλευρές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, έχουμε μόνο 16 ε, καμπίνες, συγγνώμη που δεν υπήρχαν κροατικά και ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας. Επόμενος Χωσέ Ιγνάσιο Φάρια. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κίλανεν για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και επίση να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και οι συζητητέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση των προσφύγων ε, δεν έχει προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος κύριος ε, Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στην ομιλία του για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολήθηκε με το θέμα αυτό για 45 περίπου λεπτά. Ορισμένα κρατημέλη ανέστηλαν τη συμμετοχή τους στο Σέγκεν. Η κατάσταση στην Ευρώπη είναι περίπλοκη και μοιάζει να μην υπάρχει αλληλεγγύη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να βρει μια λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ευρωπαϊκή κοινότητα γιατί είναι απαραίτητο να επιδεικνύουμε αλληλεγγύη εξετάζουμε το θέμα των ετούντων άσυλων, των προσφύγων, των μεταναστών. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα ξανασκεφτούμε και νομίζω στην Επιτροπή Μεταφορών πρέπει να εξετάσουμε τα εξή σημεία. Πρώτον, πρέπει να καθίσταται απόλυτα σαφές το ε, ποιος είναι ο τελικός στόχος ε, αυτής της έκθεσης. Οι ευρωπαϊκοί φορείς είναι εκείνοι που οργανώνουν την αντίδρασή μας στην κρίση. Η Frontex, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασύλου. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να προβληθούν περισσότερο. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο είναι, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, τα εμπορικά σκάφη είναι δέσμευσή μας να προσφέρουμε βοήθεια ε, σε όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα άλλα. Υπάρχει και σχετική συνθήκη. Η διάσωση ανθρώπινων ζώων είναι το πρωταρχικό μέλημα όλων και πρέπει να είναι και κατόπιν τούτου οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εκμετάλλευση των ιδιωτικών σκαφών. Άλλα σκάφη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τέτοιους σκοπούς και όχι ε, εκμετάλλευση κάποιων ιδιωτικών σκαφών. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι τα ιδιωτικά σκάφη απλά δεν είναι προετοιμασμένα και εξοπλισμένα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχουν αρκετούς ε, γιατρούς παραδείγματος χάρη. Οφείλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των σκαφών θα εξαναγκαστούν να ε, εξοπλίσουν σωστά αυτά τα σκάφη με δικά τους έξοδα. Επίσης, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε αναπτύσσονται τέτοιου είδου δραστηριότητε θα επικρατεί πάντα η καλή πίστη. Θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς ε, που ασχολούνται με την ασφάλεια. Σημασία έχει να ε, σώζουμε ζωές. Είναι λοιπόν μεγάλη σημασία να ενισχύσουμε τη δυνατότητά μας να συνδράμουμε σκάφη στη Μεσόγειο και επίση αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει καλύτερη συνεργασία τόσο σε θέματα ασύλου όσο και όσον αφορά τους πρόσφυγες. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δύσκολο να μην τον αγγίζει κανείς αυτό το θέμα, παρά το γεγονός ότι πιστεύω ότι ε, στο τέλος ε, η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας θα έπρεπε να αφορά κυρίως τα θέματα των μεταφορών. Είναι πάντοτε μεγάλος πειρασμός να διευρύνουμε βέβαια τη συζήτηση και το πεδίο της γνωμοδότησης αυτής. Ε, η ΑΦΕΤ και η ΛΥΜΠΕ έχουν μια κοινή συνεδρία για το θέμα αυτό και δικαίως όλοι το συζητούν. Είναι πραγματικά μια μια κατάσταση που θα δοκιμάσει την Ένωση. Είναι ε, το θέμα της αλληλεγγύης που διακυβεύεται και είναι κάτι που πρέπει όλοι να συνδυτοποιήσουμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τίμημα ανθρώπινες ζωές. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα συζήτησης. Όμως ε, εδώ συζητούμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών, οπότε ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε και σε αυτά. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της, επειδή έθεσε τα θέματα και μπορούμε να υποστηρίξουμε τα περισσότερα από αυτά. Το σημείο 7 ε, θα καταθέσουμε τροπολογία, γιατί η εισηγήτρια εδώ ζητά ε, προ, αύξηση των κονδυλίων για τις ε, προσωρινές ε, επιχειρήσεις διάσωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε αυτές οι επιχειρήσεις διάσωσης ε, να είναι μόνιμες, ότι θα έπρεπε να είναι μόνιμη υποστήριξη για αυτές τις επιχειρήσεις. Γι' αυτό Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει το σημείο προ αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι η εστίασή μα θα πρέπει να είναι στην ασφάλεια. Η ασφάλεια των προσφύγων που ε, ταξιδεύουν στην Ευρώπη, των ομάδων διάσωση, ε, αλλά και ο πολύ σκιώδη εισηγητέ το ανέφεραν αυτό, ε, τα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία μερικέ φορέ συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Δεν μπορείτε να τα υποχρεώσετε να βοηθήσουν, αλλά βέβαια θα υπάρξουν πάντοτε ε, πάντοτε μπορεί να βρεθεί κανείς σε μια κατάσταση κατά την οποία θα χρειαστεί να βοηθήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν τα ιδιωτικά σκάφη να αποζημιώνονται για την ενδεχόμενη ζημία που θα τους προκληθεί. Γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι δεν θα έπρεπε να ε, βοηθήσουν γιατί μπορεί να ε, υποστούν ζημίες για τις οποίες δεν θα αποζημιωθούν. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Οποιοςδήποτε βρίσκεται στη Μεσόγειο και βλέπει έναν πρόσφυγα σε μια δύσκολη κατάσταση πρέπει να τον βοηθήσει και πρέπει να βελτιώσουμε τις ομάδες διασωσής μας. Χρειάζεται μια μόνιμη λύση, μόνιμη χρηματοδότηση, αλλά εάν τελικά καταλήγει να το κάνει αυτό ένα ιδιωτικό σκάφος, πρέπει να αποζημιώνεται γι' αυτό. Δεν είναι επιλογή το να μην βοηθήσει κάποιος και νομίζω ότι το να βελτιώσουμε την ασφάλεια είναι ένας από τους στόχους που μπορούμε να συμπεριλάβουμε ε, στη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, συνειδητοποιώντας βέβαια ότι αυτή η ανθρώπινη τραγωδία δυστυχώς δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα. Grazie Presidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι και σε αυτή την Επιτροπή έχουμε να κάνουμε με το πρόβλημα της μετανάστευσης. Είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αυτή η πρόκληση, γιατί πράγματι πρόκειται για μια ε, ουσιαστική πρόκληση. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα, όπως έχω ακούσει να το λένε πολλοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο. Αρκετές φορές ε, χρησιμοποιείται η λέξη μετανάστευση και σε σχέση με την διασυνοριακή εγκληματικότητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, ακόμα και εδώ το θέμα δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα 500 εκατομμύρια πολίτες ε, όπου ανάμεσα αυτούς έχουμε και πολίτες εκβιομηχανισμένων κρατών ε, ότι έχουν δεχτεί κάποιες χιλιάδες ε, μετανάστες που αυτοί όμως ξεφεύγουν από τον πόλεμο και την πείνα. Το πρόβλημα είναι η πολιτική που εφαρμόζεται. Οι συνέπειες αυτών των πολιτικών ε, γίνονται αισθητέ και σε άλλες, άλλους τομείς, ε, μακροοικονομικούς ή και στις μεταφορές. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η συνάδελφος αναφέρει τον αριθμό των μεταναστών που μέχρι τώρα έχουν γίνει αποδεκτοί στην Ευρώπη. Πρέπει να το πούμε, μερικοί αποβιβάζονται, πολλοί εξ αυτών στις ε, ακτές της Μεσογείου, κυρίως στις Ιταλικές. Χαίρομαι λοιπόν που εκφράζεται για την ατελή προετοιμασία των σκαφών και του προσωπικού, γιατί πραγματικά υπάρχει κίνδυνος να χαθούν πολλές ε, ζωές. Η έκθεση λοιπόν πολύ σωστά ε, εκφράζει την άποψη της Επιτροπής Μεταφορών και κάνει λόγο για τους μετανάστες και την απόβασή τους ε, στα, σε ασφαλές μέρος. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή αυτή με θάρρος ε, να πει πολλά περισσότερα. Ε, η Μεσόγειος είναι κατά κύριο λόγο ο χώρος όπου μετακινούνται οι μετανάστες και θέλουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει να ε, μην υπάρχουν πια θάνατοι στη θάλασσα. Ζητώ καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες και όχι μόνο της Μεσογείου. Και γενικότερα μια εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο περιεκτική και να ε, βάζει ως πρώτη προτεραιότητα τις μεταναστευτικές ροές. Ε, θέλουμε καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών ανάμεσα στα 28 κράτη. Αρκεί πια το να μιλάει κανείς για όλα αυτά σε όλες τις επιτροπές, αλλά τελικά το πρόβλημα να μην λύνεται. Πρέπει να επιληθεί και μπορεί να επιληθεί εφόσον υπάρχει η πολιτική βούληση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαρή Κριστίνα Νότου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Όμως εμένα με εξέπληξαν κάποια επίθετα που χρησιμοποιήσατε. Είπατε στην αρχή ε, εθνικιστικές ε, κάποιες ε, κυβερνήσεις ή πολιτικές ομάδες που ήθελαν να προστατεύσουν κάπως τους συμπολίτε τους ανεξαρτήτως προέλευσής τους. Τέσσερα εκατομμύρια άστεγους έχουμε και περίπου 6 εκατομμύρια άνεργους. Θα έφερα λοιπόν να σας πω το εξής για όλους μας είναι συναισθηματικό το ζήτημα, αλλά δεν πρέπει πάντοτε να αντιδρούμε συναισθηματικά. Τι θα προσφέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτούς τους μετανάστες. Τι στέγη, τι δουλειά, τι είδους ε, ε, ζωή, γιατί εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών και για ποιο λόγο πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, το λαθρεμπόριο και τη λαθρέα είσοδο στις χώρες μας. Αυτό που ζούμε σήμερα ε, δεν είναι καινούριο. 10-12 χρόνια ε, ζούμε ε, το να υπάρχουν πτώματα της Μεσογείου στη Λαμπεντούζα υπήρξαν πολιτικές οι οποίες ήταν καταστροφικές και σε μεγάλο βαθμό ήταν καθαρά οικονομικές ε, γιατί πολλές φορές αν ανοίξαμε το, τα σύνορα τόσο πολύ ήταν για να μειώσουμε το κόστος εργασίας διάφορες χώρες της Ένωσης και να μειώσουμε και τις θέσεις απασχόλησης τελικά. Ε, βρεθήκαμε και το γνωρίζει και η Γερμανία της ε, κυρίας Μέρκελ με πολύ ε, ε εργατικό δυναμικό μεταναστών, ε, με χαμηλού ε, ε, μισθούς, το γνωρίζετε πολύ καλά. Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτό το μεταναστευτικό κύμα, πώς θα το διαχειριστούμε, εγώ νομίζω και ξέρω ότι δεν θα τη βρούμε τη λύση εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά εάν δεν σκεφτούμε διαφορετικά, δηλαδή να πούμε ότι να δούμε τι θα κάνουμε στις χώρες τις οποίες αποσταθεροποίησε η Ένωση και το ξέρω ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας και κυρίως οι προηγούμενες κυβερνήσεις ε, τη Λιβύη και άλλες χώρες αποσταθεροποίησαν με αποτέλεσμα αυτά που βλέπουμε σήμερα. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες αυτές γιατί δεν νομίζω σε καμία περίπτωση εγώ τουλάχιστον ότι αυτοί οι καημένοι άνθρωποι που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι προσπαθώντας το. Ε, να τους βοηθήσουμε να επιβιώσουν στις χώρες τους, να μείνουν στις χώρες τους, να δουλέψουν στις χώρες τους. Προφανώς χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική συνεργασία για να το πετύχουμε αυτό. Νομίζω όμως ότι εάν επιμείνουμε σε αυτήν την υποδοχή μιας μετανάστευσης ε, ε, που θα πλημμυρίσει την Ευρώπη, νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στις χώρες μας που θα πρέπει να τα διαχειριστούμε και είναι δική μας ευθύνη να τα αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Κριστίν Χοβοντολόν. Θα αλλάξω λίγο τόνο σε σχέση με την προλαλή σας. Η διάσωση στη θάλασσα ενό ανθρώπου που κινδυνεύει είναι ηθικό καθήκον και διεθνής υποχρέωση και τα εμπορικά σκάφη εξακολουθούν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο. Ωστόσο τα σκάφη αυτά δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να χρησιμοποιούνται σε τέτοια κλίμακα ε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, κινδυνεύουν να υφίστανται και κυρώσεις και πρόστιμα ε, όταν μεταφέρουν επιβάτες που δεν είναι, είναι παράτυποι μετανάστες. Ορισμένα σκάφη αρχίζουν να αλλάζουν δρομολόγια για να μην πέφτουν πάνω στα σκάφη των διακινητών και διστάζουν όλο και περισσότερο να δημοσιοποιούν το στίγμα του στη θάλασσα. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν ε, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ευρείας κλίμακας επιβάλλεται και δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των ε, ε, μεταφορέων που για λόγους ανθρωπιστικούς βοηθούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όπως είπαμε και στο ψήφισμα που ψήφισαμε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Τα κράτη-μέλη κατά τα άλλα θα πρέπει να σκέφτονται αποζημιώσεις προς τους πλειοκτήτες για διαφυγόντα κέρδη κατά τη διάρκεια της έρευνας και διάσωσης. Έτσι δεν θα αλλάζουν δρομολόγιο και ρότα τα πλοία ε, και ε, θα κάνω σχετικές προτάσεις για να βελτιωθεί η γνωμοδότηση που είναι ήδη πάρα πολύ ισόρροπη και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Η κυρία Λουχασεύσκα. E, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τώρα πια ε, όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν το θάρρος να μιλάνε ειλικρινά για τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ε, στη δική μας την Επιτροπή μπορούμε να υιοθετήσουμε τις καλύτερες εκθέσεις, αλλά γνωρίζουμε ότι ακόμα και αυτές οι καλύτερες εκθέσεις δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Μπορούμε βεβαίως να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, αλλά στη τελική ανάλυση συμφωνώ με εκείνους που ισχυρίζονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά ε, το αγνόησε το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ευρωπαϊκοί λοιπόν θεσμοί ευθύνονται για τις απαντήσεις ε, που έχουν δοθεί ε, και πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια που λέει ότι τα κράτη λειτουργούν ε, ορμόμενα από εθνικιστικά κριτήρια. Όχι, τα κράτη λειτουργούν υπεύθυνα. Τα κράτη καλούνται να σκέπτονται τους δικούς τους τους ε, πολίτες. Και εγώ συμφωνώ με όλους εκείνους που λένε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει βοήθεια. Οφείλουμε να βοηθήσουμε εκείνους ε, που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, αλλά μην ξεχνάμε αυτοί όλοι οφείλουν να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Επίσης, οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι αυτές ε, η κατανομή αυτών των ε, κατοίκων των 100.000 ε, δεν είναι εύκολο πράγμα στην Ευρώπη και αυτό ισχύει για σήμερα. Αύριο θα έχουμε 200-300.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Η κατάσταση λοιπόν πρέπει να αναλυθεί εντελεχώς. Και οφείλουμε επίσης ε, να αναζητήσουμε και τα αίτια που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα αίτια, γιατί η κατάσταση των ε, μεταναστών είναι τόσο κακή. Ε, και υπάρχουν και δικαιολογημένοι φόβοι κρατών, αν θέλετε, γιατί υπάρχουν κράτη που δεν έζησαν ως απικίες κατά διάρκεια των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Ε, εμείς ήμασταν χρόνια ολόκληρα κλεισμένοι, ήμασταν ε, ομοιογενείς ε, πληθυσμοί και τώρα παρότι υπάρχουν προσπάθειες είναι δύσκολο να πείσει κανείς τους πολίτες να δείχνουν ανεκτικότητα. Εμείς βεβαίως ντρεπόμαστε για εκείνους που κάνουν κηρύγματα μίσους, τέτοιοι όμως άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπεται κάθε κράτος ε, να ε, λαμβάνει τις αποφάσεις του με δική του ευθύνη. Η ε, φιλοξενία και η αποδοχή των μεταναστών. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το σημαντικότερο είναι να καταρτιστούν προγράμματα έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν στην κοινωνία και να μην δημιουργείται μία παράλληλη κοινωνία. Οι άνθρωποι αυτοί ε, δεν θα πρέπει να είναι μόνο αποδέκτες ε, κοινωνικών εισφορών ε, και παράλληλα όμως να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να σας τα περιγράψω όλα αυτά. Τα ξέρετε πολύ καλά. Είναι λοιπόν πολύ καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιληφθεί του θέματος. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η συζήτηση, οφείλουμε να ζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα. Αν ήταν θα είχε λυθεί εδώ και καιρό. Θα ήθελα όμως να παραθέσω αυτά που είπε ο κύριος Γιούγκερ, που ανέφερε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Η ε, ταχεία αντίδραση της Ευρώπης σε κρίσεις, αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι το δυνατό μας σημείο. Κατόπιν τούτου το πρόβλημα ε, εντοπίστηκε εδώ και αρκετά χρόνια, το ανέφερα προηγουμένως ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, όμως η δική μας αντίδραση υπολείπεται του αναμενόμενου. Επαναλαμβάνω λοιπόν για άλλη μια φορά ότι ακόμα και τις τέλειες εκθέσεις να εκπονήσουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Οφείλουμε ε, τις δικές μας προτάσεις, να μην τις επιβάλλουμε στους άλλους, το πρόβλημα πρέπει να το αναλύσουμε στο σύνολό του με όλες τις δύσκολες πτυχές του και δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι το να δεχτεί κανείς πρόσφυγες λύνεται το πρόβλημα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Λουντ Γκριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή τη δύσκολη κατάσταση τη βιώνουμε στη Μεσόγειο. Πάρα πολλοί καταβάλουν μέχρι και 10.000 δολάρια σε διακινητές και αυτοί, αυτούς τους φορτών τους κακόμιλους ανθρώπους ε, πάνω σε κάραβα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, πρέπει να εκπονήσουμε και τα σωστά μηνύματα. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα θέματα δεν τα εξετάσαμε σωστά. Και βλέπουμε ποιες ήταν οι συνέπειες. Ξέρετε τι κάναμε εμείς ε, ασχολιάμασταν μόνο με το αποτέλεσμα και όχι με τα αίτια του προβλήματος. Μιλάμε τώρα για 60.000 ανθρώπους και τέτοιου είδου ε, ροές μεταναστών δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να παραμείνουν στις πατρίδες τους, ε, να ζήσουν εκεί, να τους ε, βελτιώσουμε τις υποδομές, τις κατοικίες, την παροχή πόσμου νερού. Παραδείγματος χάρη στηρίζουμε τη Σομαλία. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα και προσπαθούμε εκεί να δημιουργήσουμε μια δημοκρατική κοινωνία, να προσφέρουμε τις υποδομές έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν κανένα λόγο να εγκαταλείψουν τη χώρα του, αντίον ε, να αποφασίζουν οι άνθρωποι να μείνουν εκεί. Στην ε, Σομαλία που επισκέφτηκα πρόσφατα, καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες που σας είπα Παναλαμβάνω αυτό που έχει σημασία είναι να αναζητούμε τα αίτια και όχι τις συνέπειες. Αυτό είναι πρόκληση για μένα και για μένα η πρόκληση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται λύση. Δεν ε, έχουμε βρει καμία λύση, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν είναι απλά να συνεχίσουμε διακατάσταση. Το θέμα δεν είναι να σβήνουμε κάποιες ε, πυρκαγιές, το θέμα είναι να σβήσουμε όλες τις πυρκαγιές και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχουν σειράξεις και οι άνθρωποι αυτοί να παραμένουν στις πατρίδες τους. Τα σκάφη να αναχαιτίζονται πριν έρχονται. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική για το προσφυγικό που να είναι λογική. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Έχω άλλους τέσσερις που έχουν ζήσει το λόγο αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο γι' αυτό παρακαλώ να είσαι σύντομη. Ο κ. Βαντεγκάμπ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ πάρα πολύ καλά ότι η συζήτηση ε, αυτή ε, καλή να συζητήσουμε γενικότερα για το πρόβλημα του ασύλου. Όπως είπε η συνάδελφος Λουκασέφσκα τώρα, ε, καταλάβαμε πώς έχει κατάσταση στην Πολωνία και τα λέει αυτά από καρδιάς. Εγώ έχω εργαστεί πάρα πολύ καιρό στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για να έχω και τη δυνατότητα να βάζω ε, και άλλες παραμέτρους Εγώ έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση για αυτά που λέει η συγγήτρια, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα αίτια όλων αυτών. Ε, θα, θα πούμε τίποτα για τη Frontex, θα πει τίποτα η, η συγγήτρια. Ε, πόσα είναι τα εμπορικά σκάφη που χρησιμοποιούνται. Ακούσαμε ότι αλλάζουν ρότα, ε, ότι υπάρχουν προβλήματα. Ε, και πολλά προβλήματα προκαλούνται από διακινητές για να μην μιλήσω για την κατάσταση στις διάφορες χώρες. Αυτή είναι η σημαντικότερη ερώτησή μου. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ε, αλληλεγγύη και για βοήθεια, τα οποία όλα αυτά κατανοώ και ξέρουμε και όλες τις δραματικές και τραγικές εικόνες που βλέπουμε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Μεταφορών, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ασχοληθεί και με τα αίτια του κακού. Δεν είναι καλή λύση να λύνεις μόνο το τελικό πρόβλημα, όπως λέμε στα Ολλανδικά. Ξέρω ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά ε, και στη Μεσόγειο πρέπει να ασχοληθούμε με τη ρίζα του κακού, με, όχι το τελευταίο φαινόμενο του. Ευχαριστώ. Ζήλε. Ε, ε, ναι, ευχαριστώ. Δεν ε, θα μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τα μεγάλα αυτά θέματα, γιατί εμείς είμαστε Επιτροπή Μεταφορών, δεν είμαστε Επιτροπή Εξωτερικών ε, Θεμάτων. Ε, πρέπει να διαφωνήσω πάντως με κάποιους συναδέλφους. Υπόθηκε ότι υπήρξαν πάρα πολλοί κοινέ προσπάθειες πολιτικής ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνώ. Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα, τα οποία ε, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ακυρώσουμε το Δουβλίνο ή ε, χιλιάδες ανθρώπους να τους υποδεχθούμε σε μια μέρα. Ήταν διαφορετικό το βάρος ε, για τις διάφορες χώρες και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα ε, στα σύνορα ε, της ζώνης Σέγγεν, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως επίσης και στις μεταφορές εμπορευμάτων και αγαθών. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις. Γιατί αν διακοπεί η λειτουργία της Σέγγεν, αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα. Αν θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους που ετούνται άσυλο να τους μεταφέρουμε ε, με εξαναγκαστικό τρόπο θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και αναστάτωση και στους ίδιους. Πρέπει λοιπόν να ε, βρούμε λύσεις οι οποίες θα έχουν συνέπειες προβλέψιμες. Δεν πρέπει να παρακολύουμε τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να, να σκεφτούμε ασφαλείς τρόπους μεταφοράς των ετούντων άσυλο και αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το να αποφευθούν πολλοί θάνατοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παύλ Τελίτσκα. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Δύο επιλογές είναι. Πρώτον, να μπω σε λεπτομέρειες όπως έκαναν πολλοί εξέχονται συνάδελφοι αναλύοντας την κατάσταση και μπαίνοντα σε λεπτομέρειες ε, για μέτρα, ε, μιλώντας για αλληλεγγύη κλπ. Πιστεύω ότι θα ανέλεια τις προτάσεις ε, της Επιτροπής με τέτοιο τρόπο ώστε να ε, δείχνει ότι είναι ανεπαρκή σε σχέση με τις αιτίε, αλλά είναι και ανεπαρκή και ως προς τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είμαστε όμως στην Επιτροπή Μεταφορών και πρέπει να ασχοληθούμε με τις συνέπειες για τις μεταφορές, για θέματα που έχουν σχέση με τις μεταφορές ε, και ε, να αφήσουμε τα υπόλοιπα για το Frontex. Τι μπορούμε εμείς να στείλουμε ως, ισχυρή, ε, ως ισχυρό ε, μήνυμα ότι αυτές είναι οι συνέπειες και αυτό πρέπει να γίνει και την πολιτική συζήτηση να την αφήσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για παράδειγμα και εμείς θα έχουμε και την ευκαιρία και στην Ολομέλεια να το συζητήσουμε αλλά τώρα χάνουμε την ευκαιρία να δούμε την πτυχή των μεταφορών όλου αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω γενικώ εγώ ότι για μένα είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Και αυτό το προσφυγικό πρέπει να λυθεί ε, στην Ευρώπη, στο σύνολό της. Αλλιώς θα καταρρεύσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα γενικά. Και καλούνται όλοι. Και η πρόταση του Τόναλτ Τούσκ ήταν καταπληκτική, διότι είπε και τα 28 κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν. Βεβαίω λαμβάνουμε υπόψη τον πληθυσμό, αλλά και την οικονομική δυνατότητα κάθε χώρα. Και βάσει αυτών έκανε πρόταση. Και εκεί υπάρχουν χώρε που δεν θέλουν να συμμετέχουν. Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Θα μπορούσε ο καθένα να έχει του λόγου του. Για να επανέλθουμε λίγο στην ιστορία, μια αναδρομή τη ζήσαμε στην Ευρώπη. Εγώ είμαι από τη Γερμανία από το 59 μέχρι το 61 μέχρι να χτιστεί το τείχος 4 εκατομμύρια άνθρωποι ε, έφυγαν από την Ανατολική Γερμανία προς τη Δυτική για να γλιτώσουν και είχαμε και τους πρόσφυγες από την Πολωνία και από άλλες χώρες που ήταν Γερμανοί που ζούσαν εκεί και δεν είπαμε να φροντίσουμε να ζουν εκεί αυτοί οι άνθρωποι αλλά δείξαμε προθυμία να τους βοηθήσουμε. Όταν το 68 έγινε επανάσταση στη Τεχοσλοβακία και ε, ε, στείλανε τα τάγκς οι Σοβιετικοί πάλι έφυγαν πάρα πολλοί προς την ε, Αυστρία, Γερμανία, την Ευρώπη. Κανείς δεν είπε να μείνουν στην Τεχοσλοβακία να ζήσουν. Τους βοηθήσαμε και ε, το κάναμε αυτό. Ε, ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα. Το 1956 στην Ουγγαρία θυμάστε τι έγινε όταν κατέβηκαν τα τάγκ στην Επανάσταση. Και πάλι μέσω της Αυστρίας ήρθαν στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη που ήταν πολύ μικρότερη από τη σημερινή. τους δεχτήκαμε, για τους υποδεχτήκαμε όλους. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι η αρχή. Αυτό είναι το κεντρικό, το κομβικό ζήτημα δεν λυθεί ευρωπαϊκά, τότε θα πάει περίπατο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και η Ευρώπη δεν είναι πώς θα μοιραστούμε τα λεφτά. Έχουμε αξίες και αρχές που πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Βεβαίως και με τα αίτια. Τι κάναμε στην αναπτυξιακή πολιτική τα τελευταία 20-30 χρόνια. Μήπως ε, ε, κερδοσκόπησαν οι, οι πλούσιες χώρες αντί να βοηθήσουν. Τώρα όμως χρειάζεται βοήθεια, θα τα δούμε και τα άλλα. Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιωτικά σκάφη που θα πρέπει να τρέξουν ή τα εμπορικά πλοία να κανονίσουν την πορεία τους και ότι εκεί είναι τα ελλείμματα. Φυσικά και θα πρέπει να αποζημιώνονται. Είναι σαφές αυτό. Αλλά είναι το θέμα κεντρικό, πολιτικό, εμείς τώρα το κοιτάμε από το πρίσμα της Επιτροπής Μεταφορών. Είδαμε στη Σύραγγα, στη Μάχη, στο Καλέ τι γίνεται και θα πρέπει να κάνουμε προτάσεις και γι' αυτό. Γενικά πιστεύω όμως είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Αρκεί να σκεφτώ. Ε, σε 12 χρόνια, από το 49 μέχρι το 61, τα 4 εκατομμύρια ε, που ήρθαν από την Ανατολική Γερμανία στη Δυτική, σημερινά νούμερα είναι μικρά. Ε, Πάντω η λύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Α, puheenjohtaja. Hyvät arvostetut. πολύ. Α, ευχαριστούμε πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Με βάση λοιπόν αυτή τη συζήτηση κατέληξα στα εξής ε, συμπεράσματα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας ε, στην αίθουσα αυτή που να επιθυμεί να στηριχθεί το οργανωμένο έγκλημα και η συμμορία των διακινητών. Εμείς ε, τα προβλήματα θέλουμε να τα επιλύσουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εισέρχονται νόμιμα και να μπορούν ε, να ζητήσουν έκτακτη βοήθεια. Όσον αφορά τα εμπορικά σκάφη, βεβαίως ε, όλα αυτά ε, τα κατέγραψα και κανείς δεν επιθυμεί στην Μεσόγειο να εκτροχιαστεί η κατάσταση, οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους και η φύση να εφίσταται μεγάλες ζημιές. Ούτε επιθυμεί κανεί οι διακινητέ να επιτίθενται σε ευρωπαϊκά σκάφη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές. Στόχος μας είναι να σώζονται ανθρώπινες ζωές και το βάρος πρέπει να επιμερίζεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτή όμως η ανθρώπινη διάσταση δεν πρέπει να χαθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να μας. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να βρούμε μία λύση που να ικανοποιεί όλους. Όμως ε, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα πριν κατατεθεί η έκθεση φαντάζομαι θα πάρουμε από εσάς ε, πολύ καλές ε, προτάσεις και με βάση αυτές θα μπορέσουμε ελπίζω να καταλήξουμε σε καλούς συμβασμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά ε, είχαμε μία ουσιαστική συζήτηση Είχα φανταστεί ότι ενδεχομένως να συγκρουστούμε, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ε, ευχαριστώ και τους και όδης εισηγητές και είμαι αισιόδοξη ότι τελικά θα καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό κείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Η 7η Σεπτεμβρίου είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάψη τροπολογιών. 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Είστε πάλι εσείς η συγγήτρια, η κυρία Κιλόνεν προς μια νομοθετική πράξη για την νέα ψηφιακή αγορά. Μόλις ολοκλήρωσε την προηγούμενη έκθεσή της και τώρα έχει και πάλι το λόγο. Κυρία Κιλόνεν, έχετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το καλοκαίρι προετοίμασα αυτήν ε, την έκθεση της Επιτροπής μας ε, για την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά. Καλό είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την άποψη της Επιτροπής ε, του, του κλάδου των μεταφορών ε, για το σημαντικότατο αυτό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως προτείνει ε, μέτρα τα οποία είναι κάπως περιορισμένα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο τομέας των μεταφορών θα επηρεαστεί πάρα πολύ από την ψηφιοποίηση σε όλο τον κόσμο. Θα υπάρξουν πάρα πολλές συνέπειες. Πρώτον, οι χρήστες, οι πελάτες, όλο και περισσότερο δραστήριοι θα είναι στο πλαίσιο του συστήματος μεταφορών. Δεύτερον, οι πληροφόρηση, ενημέρωση θα είναι όλο και σημαντικότερη γιατί θα υπάρξουν νέα μοντέλα επιχειρήσεων ε, και βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ε, όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένοι, ε, είναι όλο και περισσότερο ψηφιοποιημένος και ο διάλογος μεταξύ των πολιτών. Θα ήθελα να μπω σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες τώρα. Αυτά ήταν τα γενικά μου σχόλια όσον αφορά στους χρήστες και τους πελάτες όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο ενεργοί θα είναι, λιγότερο παθητικοί, λιγότερο άδρανοι, θα έχουν όλο και περισσότερο τη ε, δυνατότητα να ε, διαλέξουν, να σχεδιάσουν τον τρόπο της μεταφοράς τους. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι παροχής πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο τρόπο μεταφορών. Η πληροφορία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι όλο και σημαντικότερη. Αν δεν κυκλοφορεί η πληροφορία δεν κυκλοφορεί τίποτα. Είναι κατά κάποιο τρόπο το πέμπτο είδος μεταφορών σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ε, τα κενά ενός ταξιδιού αν για παράδειγμα κάποιο περιμένει στη στάση του λεωφορείου, προτιμά να έχει ακριβεί πληροφορίες από το να έχει μεγαλύτερη συχνότητα ε, λεωφορείων. Αυτό σημαίνει ότι οι καλύτερες πληροφορίες ενημερωμένες ε, για τους ε, πελάτες είναι φθηνότερο από το να βάλει κανείς σε κυκλοφορία περισσότερα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη υπάρχει το θέμα της προστασίας των δεδομένων και της εμπιστευτικότητας που είναι στο επίκεντρο αυτής της ε, ενιαίας αγοράς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν τα αυστηρότερα μέτρα, αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών και να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων. Χρειαζόμαστε υποδομές ε, ε, δεδομένων λειτουργικές, διαλειτουργικές και διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων χωρίς κανένα, καμία ανεπάρκεια και χωρίς κανένα κενό από απόψεως ασφαλείας. Υπάρχουν νέα ε, μοντέλα ε, και στον κλάδο των μεταφορών κατά τα επόμενα έτη θα αλλάξει άρδιν ε, ο τομέας των μεταφορών και θα χρειαστεί να αλλάξει όπως έγινε και στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα του τουρισμού προσφάτως. Προφανώς ε, θα υπάρξουν πάρα πολλά ε, ωφέλη για τις ε, μεταφορές με την ύπαρξη νέων φορέων. Google για παράδειγμα, η οποία αναπτύσσει συστήματα πλοήγησης αυτόματα. Εκτός από τους παραδοσιακούς παίκτες, τους διαχειριστές υποδομών, επιμελητίας, τις μεταφορές, τα ταξί, υπάρχουν και νέοι παίκτες παίκτες ε, που διαφαίνονται. Υπάρχουν οι διαχειριστές των υπηρεσιών που συνδέουν τα, τους νέους τρόπους μεταφορών με τους πιο παραδοσιακούς. Το ίδιο ισχύει και για αυτό που λέμε τώρα νέα τεχνική ανταλλαγής. Υπήρχαν κάποια φαινόμενα αρνητικά, όμως κατά γενικό κανόνα και μιλάω για, τους, ε, τα νέα ε, είδη, τους νέους τρόπους μεταφορών ε, που είναι φθηνότερα, πιο εύκολα για τον καταναλωτή και ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του. Πρέπει να δούμε λοιπόν την έμεση αξία της, των μεταφορών, πώς μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τελικού χρήστη, Είτε πρόκειται για έναν ιδιότητα, είτε πρόκειται για κάποιον που μεταφέρει εμπορεύματα η ψηφιοποίηση ε, στον τομέα των μεταφορών ε, ανοίγει τεράστιο δυναμικό αύξηση των θέσεων απασχόλησης, οι οποίες αυτή τη στιγμή μας λείπουν, τις χρειαζόμαστε. Η ανάπτυξη του, ε, των εφιών μεταφορών είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πάνω από 16% είναι κατά την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη του και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. το διαδίκτυο των πάντων ε, θα μπορούσαμε να πούμε πλέον. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για όλα. Και στο τομέα των μεταφερών όλο και περισσότερες εφαρμογές θα μπορούσαμε να είχαμε ε, για αυτού του είδους το διαδίκτυο να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, οχημάτων για παράδειγμα υποδομές ε, με μετακίνηση πολύ πιο ρευστή και πολύ πιο σίγουρη ανταλλαγή πληροφοριών πάρα πολύ γρήγορη είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι πώς μπορούμε να αντιδράσουμε Κατά την άποψή μου, η ψηφιοποίηση είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα σύστημα μεταφορών ακόμη πιο αποτελεσματικό, ακόμη πιο παραγωγικό, με ε, μια επιμελητία πιο ρευστή, πιο αποτελεσματική, λιγότε, που είναι λιγότερο δαπανηρή και σέβεται περισσότερο την οικολογία. Τώρα πρέπει όμως να υπάρξει το απαραίτητο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό. Και προτείνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μία αξιολόγηση ως προς τις ανάγκες εναρμόνισης των κανόνων των διαφόρων τρόπων μεταφορών για να υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων ε, τρόπων μεταφορών και μπορούμε έτσι να προωθήσουμε υπηρεσίες ε, καινοτόμες. Δεν χρειάζεται όμως να μπαίνουμε και δεν χρειάζεται όμως να ε, ε, υπάρχουν κακές συνέπειες ε, σε θέματα όπως η προστασία των καταναλωτών, δεν πρέπει να, υπάρξει, να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον. Αντιθέτως πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε κάθε ε, φορέας να μπορεί να αξιοποιήσει αυτήν τη νέα κατάσταση και να την εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Πάντοτε όμως δεν πρέπει, ποτέ όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει αυτή η έννοια των αναγκών των καταναλωτών. Οπότε θα γίνουν τροπολογίες λαμβάνοντας, ε, θα λάβουν υπόψη τη διατροπικότητα, τα δικαιώματα των επιβατών, ε, την έκδοση εισιτηρίων, το σύστημα πληροφόρησης. Αυτές τις ε, προτάσεις, αυτές τις τροπολογίες θα τις συζητήσω με τους σκιώδεις εισηγητές. Μπορείτε να τις υποστηρίξετε ή να τις απορρίψετε. Και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω το εξής. Ανέφερα σημαντικά σημεία που για μένα ε, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη, δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με την ψηφιοποίηση κλπ. Θα ήθελα όμως, αν σας ενδιαφέρει, να σας καλέσω στις 14 Οκτωβρίου σε μία ακρόαση το πρωί. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά ε, με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων θα σας στείλω και ένα email σχετικά με την ακρόαση αυτή. Και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, αν θέλετε, να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, των μεταφορών και της ψηφιοποίησης λεπτομερέστερα. Ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων των τον, των, ε, σκιώδης για τις παρατηρήσεις τους ε, που μου επέτρεψαν ε, να καταλήξω στο πρώτο αυτό έγγραφο. Αναμένω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε κλον. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και για τις προτάσεις της και για την έκθεσή της. Είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο ε, ως πλατφόρμα για να συζητήσουμε τις διάφορες προσκλήσεις της ψηφιοποίησης στο τομέα των μεταφορών. Και η έκθεση για το ενιαίο εισιτήριο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και εστιάζει και καταδεικνύει πόσο μπορεί να βοηθήσει η ψηφιοποίηση ε, ε, τους επιβάτες για την τιμολόγηση, για την ε, ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα τρένα και όλα αυτά, για, τα, για όλες τις μεταφορές. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τις εμπορευματικές μεταφορές, οδικές, πλωτές, ποτάμιες, τα κτλ. Υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας για μεταφορείς, για χρήστες, για βελτιστοποίηση. Ε, μπορούν να δουν ε, τι ε, δρόμους θα χρησιμοποιήσουν, τι βιγές, τι... Είναι τεράστιο το δυναμικό για την καλύτερη διαχείριση και την επιμελητία γενικά στην εφοδιαστική και όπως λέει και η ήτρια μπορεί να προβλέψει κανείς καθυστερήσεις λόγω επεισοδίων ή λόγω δυστυχημάτων, να κάνει παράκαμψη και να κερδίσει χρόνο κτλ. Ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά χρειάζονται και τα έγγραφα για να έχουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών. Το ξέρω, το ακούω αυτό το επιχείρημα που λέει ότι εντάξει δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε και πάρα πολλά έγγραφα και τέτοια γιατί υπάρχει ένα θέμα προστασίας. Αλλά ε, ε, ρωτάς κάποιον που είναι οι αποθήκη σου, ε, ποια είναι η ε, εφοδιαστική σου κτλ. Και, και πρέπει να σου αποκαλύψει όλα τα στοιχεία της επιχείρηση είναι ένα ζήτημα. Από πλευράς ε, μεταφορών, ε, από τη δική μας σκοπιά, πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε και να κάνουμε. Τα είπε και η συγγήτρια και τα περιέγραψε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουμε ε, ένα ενιαίο διαβιβαστικό κείμενο Ε, ε, να έχουν ενιαία έγγραφα, εν πάση περιπτώσει, ή μεταφορείς. Ε, Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή και στεναρή έκθεση για να τονίσουμε και τη σημασία όλων αυτών. Ευχαριστώ η Όλγα Σελάνοβα. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τοποθέτησή σας, και επίσης την ευχαριστώ πάρα πολύ και για την προτιμία που επέδειξε να συνεργαστεί με τους και ηγητές σε αυτή τη φάση. Εμείς πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή και ε, λαμβάνει υπόψη της ε, τις νέες δυνατότητες ε, που υπάρχουν, τη νέα τεχνολογία. Η συγγήτρια λέει ότι ο ρόλος κλειδί στην ψηφιακή αγορά είναι η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων. Και αυτό από κοινού με την τεχνολογία και τη διαλειτουργικότητα, αυτό θα συμβάλλει σε μια καλύτερη κατάσταση στην Ευρώπη. Βεβαίω μπορεί κανεί ε, να λειτουργήσει προληπτικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να συμβάλλει. Εξάλλου ε, το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και ορισμένα σημαντικά στοιχεία της ασφάλειας, της διασφάλισης των ε, θέσεων εργασία και της προστασία του καταναλωτή. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το σημείο εκείνο όπου αναφέρεται ότι η προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Ε, βεβαίως η γνωμοδότηση δεν είναι αρκετά περιεκτική. Εμείς ε, θα θέλαμε ευχαρίστως ε, τη γνωμοδότηση αυτή να την διευρύνουμε κατά για να υπάρχουν λεπτομερέστερες περιγραφές. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω δύο πράγματα. Πρώτον, τα νέα ICT θα πρέπει να είναι πιο προσπελάσιμα για όλους τους πολίτες. Και αυτό αφορά και πολίτες ε, που έχουν ε, κάποια προβλήματα, είτε υποφέρουν ε, από ναυτία, είτε οτιδήποτε άλλο. Και το geo-blocking και αυτό δεν πρέπει να παρεμβαίνει, γιατί και αυτό παρεμποδίζει πολίτες να χρησιμοποιούν αυτή την εφαρμογή. Αυτές θα είναι περίπου οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε, αλλά σας λέω για άλλη μια φορά, επίσης εξ αρχής, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Κοσματολοφσκή, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Όσον αφορά τις μεταφορές, η ψηφιοποίηση είναι και μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη πρόκληση. Υπάρχουν νέες μορφές ε, παροχής ε, υπηρεσιών μεταφορών οι οποίες στηρίζονται από τις νέες τεχνολογίες και με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης ή ε, τιμές πέφτουν αλλά οι παλιές θέσεις εργασίας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχουν διαμαρτυρίες. Δεν πρέπει να έχουμε κατά νου μόνο την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ασφάλεια των επιβατών και τα φορολογικά θέματα. Ε, σε αυτά λοιπόν τα θέματα δεν θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά πρόθυμοι για συμβιβασμούς. Η ψηφιοποίηση της αγοράς ε, σημαίνει ότι θα πρέπει ε, να την χάνουν επεξεργασία σε πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια. Εξάλλου ε, πρέπει ε, να βρεθούν λύσεις για το geo-blocking, έτσι ώστε να υπάρχει και καλή χρήση των ψηφιακών ε, δυνατοτήτων. Ε, ο γεωγραφικός αποκλεισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό αφορά κυρίως ε, ανθρώπους που βρίσκονται εν κινήσει, ταξιδεύουν, βρίσκονται σε αεροδρόμια, συνδρομικούς σταθμούς, ξενοδοχεία, μόνο με τέτοιου είδους, με τέτοιου δυνατότητες μπορούμε να θεωρούμε ότι η στρατηγική αυτή θα είναι αποτελεσματική. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών στοιχείων ε, απαιτεί και προποθέτει κάποιες ικανότητες να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά τα ψηφιακά στοιχεία. Η χρήση εφαρμογών που ε, βοηθούν στο να αγοράσει κανείς ας πούμε εισιτήρια θα πρέπει να είναι εύκολη και από γλωσσικής πλευράς οι ψηφιακές ε, ικανότητες είναι πολύ σημαντικές και για την εκπαίδευση οδηγών και όλων εκείνων που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ε, βελτιώσουμε την ασφάλεια στις μεταφορές και να δημιουργήσουμε και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πάμε τέλειτσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και πρέπει να πω ότι το σχέδιο ε, έκθεσης απαντά στι ε, προσδοκίες μας και τα εισαγωγικά της σχόλια ενδιαφέροντα τα βρήκα. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για τις μεταφορές με την ψηφιακή αγορά για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Συμφωνώ. Όλο μιλάμε για αυτά τα θέματα, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεταφορές είναι από τις προτεραιότητες όλων αυτών. Και τώρα βλέπουμε ε, να συμβαίνει. Και υπάρχει μεγάλο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο για γνήσιο ανταγωνισμό. Ε, και μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς και όλων των φορέων, νέων, παλιών και να ενθαρρύνουμε φυσικά και την καινοτομία. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι ένας τομέας όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη και να μένουν εκεί και στις μεταφορές επίσης προσφέρεται ο κλάδος. Ένα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω και συμφωνώ με την εισηγήτρια είναι η σημασία να εξασφαλίσουμε ε, ε, πολύ καλή προστασία των προσωπικών δεδομένων ή ε, το δεδομένων γενικότερα. Για την ομάδα μας αυτό είναι προτεραιότητα, το ξέρετε. Συχνά λέμε ότι μπορούμε να είμαστε ηγέτης ως Ευρώπη σε πιο κλάδο της οικονομίας για τις μεταφορές. Το πιστεύω αυτό πραγματικά. Ε, και όταν το συνδέσουμε με την ψηφιακή αγορά ακόμα περισσότερο. Ε, ο τουρισμός επίσης δεν αποτελεί εξαίρεση και θα πρέπει να το λέει και το σχέδιο της έκθεση αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πάρα πολλές ανάγκες. Η δική μας ομάδα έχει εντοπίσει τέσσερις βασικούς τομείς για την ψηφιοποίηση ε, ε, πρώτα θα πρέπει να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, πάρα πολύ ωραία το λέει η συγγήτρια αυτό, ε, να αγκαλιάζουμε και καλοδεχόμαστε τις αλλαγές και να δράτουμε τις ευκαιρίες. Ίσως κάνω κάποιες τροπολογίες εδώ για το δεύτερο αυτό με τις αλλαγές και τις ευκαιρίες, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και να, να δεχτούμε ότι ο τουρισμός και ε, οι μεταφορές ε, παρέχουν, ε, πώς να το πω, ελπίδα για ένα νέο είδος κοινωνίας, ένα νέο μοντέλο κοινωνίας και οικονομίας. Αναλαμβάνουν τα ενία, οι καταναλωτές λένε τι χρειάζονται και πώς θέλουν να το επιτύχουν αυτό. Καμιά φορά οι ίδιοι οι καταναλωτές γίνονται πάροχοι υπηρεσιών. Αυτή είναι η οικονομία η συμμετοχική και η οικονομία με βάση τη ζήτηση. Στις ευκαιρίες θα πρέπει να δράξουμε επίσης. Θα πρέπει οι εταιρείε και οι καταναλωτέ να υποφεληθούν από την ψηφιακή αγορά. Αν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα έχουμε πετύχει. Είναι ένα τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία και αλλάζει και χρειάζεται ένα αριθμιστικό πλαίσιο για να υποστηριχθούν οι εταιρείε να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είτε είναι ε, με το ITS, το ενιαίο εισιτήριο, την ε, επιγραμμική προώθηση, διαφήμιση, διάφορες επενδύσεις χρειάζονται εκεί και αυτό θέλω να το τονίσω επίσης. Και αυτό είναι ένα θέμα άντλησης κοινοτικών κονδυλίων. Ξέρω ότι το έχουμε υπόψη μας και έχουμε εστιάσει σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμα μεγάλο έδαφος να καλυφθεί. Το είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση ότι θέλω να ενισχύονται όχι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά οι startups, οι πραγματικές νεοφύης. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, τη συγχαίρω, πάει σωστή κατεύθυνση και με χαρά να συνεργαστούμε. Θα φέρω και μερικές τροπολογίες για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ, η Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για ε, όλα αυτά που μας είπατε που ε, ανοίγουν τη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι η ψηφιοποίηση εκτός από τις χρήσεις καθημερινής ζωής ε, των συμπολιτών μας είναι πραγματικά κάτι που επηρεάζει την κοινωνία μας σε όλους τους τομείς της και εμείς ως πολιτικοί δεν έχουμε το ρόλο να πούμε αν η τεχνολογική αλλαγή είναι καλή ή όχι, αλλά να προβλέψουμε, να προετοιμάσουμε την αλλαγή αυτή και αυτός ο, αυτή η αλλαγή που επιφέρει η τεχνολογική αλλαγή να, σημειώσει, να, να σημαίνει πρόοδο οικονομική, περιβαλλοντική. Είναι κάτι το οποίο ισχύει βεβαίως και, στη, και στον τομέα των μεταφορών. Η ψηφιοποίηση και η επανάσταση αυτή ε, αναστατώνει και τον τομέα αλλά και τη συμπεριφορά των χρηστών, των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στην ε, προσπάθεια ε, της πληροφορίας που μπορούμε να έχουμε μέσω του ίντερνετ. Είναι όμως αυτό μια μεγάλη πρόκληση γιατί ε, στα μέσα μεταφορών ε, σήμερα. Ε, κάτι τέτοιο μας δίνει τη δυνατότητα πιο ρευστών μετακινήσεων. Μπορεί κανείς να δει τα δρομολόγια, να επιλέξει το εισιτήριό του. Ε, υπάρχουν υπάρχουν ε, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, κάτι το οποίο είναι καινούριο, ακόμη και για ε, την αναστάτωση της κυκλοφορίας στα ποτηλιαρίσματα και φυσικά πρέπει η προσφορά να ε, ανταποκρίνεται στη ζήτηση. Είναι και το θέμα της συνεργατικής οικονομίας. Σήμερα Μιλάμε για το συνεπιβατισμό, μιλάμε για τα ποδήλατα ε, που θα παρέχονται, ε, που θα μπορεί να τα παίρνει ο καθένας μόνος του. Αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια πρόκληση. Η επανάσταση της ψηφιοποίησης ε, πρέπει να έγινε και στο, στην αλλαγή της θεώρησής μας για το αυτοκίνητο είναι γεγονός ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί πραγματικότητα. Μιλάμε σήμερα για ε, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό πλέον. Τα... Αυτό σημαίνει ότι θα ψηφιοποιηθούν και οι δρόμοι ε, στο μέλλον. Ε, και εμείς πρέπει ως συνομοθέτες να παρέχουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο γι' αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι η ψηφιοποίηση πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα σύλληψη της ιδέας των μεταφορών, της έννοιας των μεταφορών, πώς μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό για ε, μεταφορές ε, οχημάτων πολύ πιο βιώσιμες και ε, το είπατε κι εσείς ότι πρέπει να προβλέψουμε τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ψηφιοποίησης και της συνεργατικής οικονομίας και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ε, έγινε η βασική μας, ε, το βασικό μας θέμα το θέμα του Uber για παράδειγμα, που είναι ένα πραγματικό ε, πρόβλημα που τίθεται και το άλλο θέμα είναι η προστασία των δεδομένων που σημαίνει βέβαια ε, ανησυχία και για τους μισθούς και το θέμα της προσβασιμότητας γιατί δεν πιστεύω ότι σήμερα ε, το σύστημα μας ε, είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρίες. Είναι κάτι το οποίο το ε, είπατε κι εσείς, το θέμα της διαλειτουργικότητας, της διατροπικότητας. Σήμερα όμως μιλάμε για διασύνδεση. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα ενταχθούν σε μια κοινή δυναμική. Βεβαίως να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την ανάπτυξη πλατφορμών, μπορούμε να μιλάμε για ε, ηλεκτρονικές πλατφόρμες κινητικότητας, ε, όμως χρειάζονται κάποια, κάποιες δικλίδες ασφαλείας, κάποιες εγγυήσεις. Πρέπει να μπορούν ε, και οι πολίτες να το καταλάβουν και πρέπει προλαμβάνοντας να έχουμε κάποια, κάποιο δίκτυο ασφαλείας ώστε να μην έχουμε προβλήματα που να υπερβαίνουν την κοινωνία μας αλλά και ε, εμάς ως πολιτικούς. Ευχαριστώ κύριο Ρικέ και παρακαλώ σύντομο γιατί έχουμε πρόβλημα χρόνου. Ευχαριστώ πολύ ε, την εισηγήτρια για την πληρέστατη εργασία της. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε. Θέλω να επιμείνω σε κάτι όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Όταν συζητούμε έτσι στα πλαίσια της αρμόδιας επιτροπής, ε, επί της ουσίας δηλαδή, υπάρχει μια πάρα πολύ καθυστερημένη άποψη ε, ε, τις σχέσεις ψηφιακής αγοράς με τις μεταφορές. Τι εννοώ. Σήμερα μόνο αρχίζει να αναδύεται αυτή η αίσθηση. Ε, επί πολύ καιρό το θεωρούσαν σύστημα πληροφορίας, πληροφορικής, διαχείρισης πληροφοριών. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και λειτουργικό και θα επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές στον ίδιο τον τρόπο και τη δραστηριότητα των μεταφορών, στην οικονομική δραστηριότητα και στις θέσεις εργασίας. Άκουσα για τα αυτοκίνητα χωρίς ε, οδηγό ή και αυτοκίνητα για συνεπιβάτες χωρίς οδηγό. 750.000 ε, ε, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στην Ευρώπη. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Και τα δύο τρίτα είναι μετανάστες πρώτης γενεάς. Καταλαβαίνετε τι σοβαρές και βαριές συνέπειες θα έχει και αυτό δεν το έχουν καταλάβει πάρα πολύ ακόμα οι μεταφορείς, οι ασχολούμενοι με τον κλάδο αυτό. Κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο σοβαρό. Στον κόσμο αυτό το ψηφιακό, η σημασία των μεταφορών και η σημασία να σταθεροποιηθούν ε, οι μεταφορές και οι υποδομές δεν έχει ληφθεί υπόψη καθόλου. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τις υποδομές, γι' αυτό το λέω. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι το ITS ή όλα τα συστήματα, τα αυτοκινούμενα χωρίς ε, οδηγό. Χθε συζητούσαμε για τα ντρόμου στην έκθεση της κυρίας Φώστερη, συζητούμε και για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό που ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για ε, συνδυασμένες μεταφορές, αυτο, ε, φορτηγά, βαρέα και τρένα. Είναι πολύ βαριές υποδομές δεν είναι ουδέτερα αυτά τα θέματα. Από ό,τι φαίνεται, ε, ο ψηφιακός κόσμος δεν έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον κόσμο των μεταφορών και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για ανάγκες και ε, για αναγκαιότητες που δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει η ψηφιακή αγορά. Κάποια στιγμή ε, δεν πρόκειται να ακολουθήσει η επιμελητία, όπως έλεγε ο στρατηγός Δεγκόλ. Ευχαριστώ, Ινέσα Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Έχει κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Πολύ αξιόλογη. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να καλύψει όλη την περιπλοκότητα του κλάδου. Ιστορικά θέλω να θυμίσω μόνο το εξή. Η ψηφιακή τεχνολογία στις μεταφορές είναι κάτι που μπήκε πολύ νωρίς ε, στα αεροπλάνα, στους δορυφόρους για τα αεροπλάνα, στα αυτοκίνητα, στα πλοία, στην επιμελητία, την εφοδιαστική, την αστική κινητικότητα. Τα ξέρω. Ξέρω ότι είναι πολύ νέα η συγγήτρια, αλλά να ξέρουμε λίγο και την ιστορική πορεία, να είμαστε και δίκαιοι με όλα αυτά που έχουν κάνει μεταφορές γι' αυτό. Ε, όλα αυτά τα θέματα λοιπόν και μάλιστα αυτές τις αλλαγές που γίνονται Πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και είναι μεγάλες οι προκλήσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε και σε συγκεκριμένα πράγματα. Πριν από λίγα χρόνια ε, είχαμε την πλατφόρμα Θαλής που μπορούσες ε, να βγάλει εισιτήριο για τους γερμανικούς σιδηροδρόμους και τούμπαλεν. Σήμερα που έχει εξελιχθεί η πλατφόρμα δεν μπορείς να αγοράσεις αυτό θαλή εισιτήριο για την Deutsche Bahn και να μην μπορείς στη χώρα μου γιατί θα με πιάσουν τα κλάματα αν αρχίσω να λέω για τη δική μου χώρα τι συμβαίνει εκεί. Ε, ένα παράδειγμα μόνο είναι αυτό. Και θέλω να σας πω ότι μην τρελαθούμε τώρα με το μέλλον και ξεχάσουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δύο πράγματα. Πρώτον, η ε, συμμετοχικές μεταφορές και η συνεργατική οικονομία, αλλά είδαμε τι έγινε με την Uber. Είναι ο άκρατος ξέφρενος καπιταλισμός. Συνδέεται ο πάροχος με τον καταναλωτή χωρίς κανένα πλαίσιο κανονιστικό, επιθεώρηση εργασίας, ε, όλα χαλήνοτα είναι, κανένα πλαίσιο δεν υπάρχει. Βγάζει ένας μια πλατφόρμα ψηφιακή και την πουλάει σαν να ήταν ε, ο νέος παράδεισος. Για κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για τους εργαζομένους όμως. Ε, μπράβο για τον καταναλωτή που είναι πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος και για τον πάροχο που κάνει τον κόσμο να δουλεύει. Αλλά τι γίνεται με τους επαγγελματίες του κλάδου. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αξιοποίηση. Και όλα αυτά για ε, τα οχήματα ε, τα αυτόματα ε, ηλεκτρονικά για τους χρήστες. Κοιτάξτε, ο πληθυσμός ε, γυράσκει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι. Δεν μπορούν να χειριστούν όλα αυτά τα εργαλεία που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία πλέον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και εσείς παρακαλώ δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που βρίσκομαι και σήμερα εδώ. Ε, δεν ξέρω αν θα είμαι τόσο σύντομη όσο πώς εχθές. Όπως ξέρετε η στρατηγική ε, της ψηφιοποίησης της ενιαίας αγοράς είναι ένα θέμα που αφορά πολλές ε, ε γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας δώσω πρώτα κάποιες ε, γενικότερες πληροφορίες έχουμε εξελίξεις που είναι πολύ σημαντικές για τις μεταφορές, γιατί το όλο σκεπτικό πίσω από αυτή τη στρατηγική είναι να καταλήξουμε τελικά σε οριζόντιες προτεραιότητες οι οποίες θα επιτρέψουν να αντιμετωπίζει κανείς ειδικέ ανάγκες. Γιατί και πάλι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ψηφιοποίησης ότι τώρα πλέον μιλάμε για αλληλένδεση και δεν είναι οι μεταφορές όπως ήταν πριν από 7 περίπου χρόνια. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων είναι πολύ σημαντική, εξίσου βέβαια σημαντική στις μεταφορές όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κατά τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εισάγει διαβουλεύσεις για την ε, γεωγραφική, γεωγραφικό αποκλεισμό. Τώρα πλέον μιλάμε για την ε, κοινή αγορά, για την ψηφιοποίηση της κοινωνικής αγοράς, ο γεωγραφικός αποκλεισμό εξακολουθεί να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Επίσης, όσον αφορά τις πλατφόρμες και εκεί υπάρχουν θέματα όπως είναι η αξιοπιστία των δεδομένων. Πολλά από τα θέματα που ετέθησαν από τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Εξάλλου, θα έχουμε και μια αρκετά εκτεταμένη διαδικασία όπου θα ε, περιλαμβάνονται όλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι για να διαπιστώσουμε αυτή η ομάδα των ε, άμεσα εμπλεκομένων πόσο ευρεία είναι η ομάδα αυτή. Δεν περιλαμβάνονται μόνο οι χρήστες και οι φορείς εκμετάλλευσης αλλά και πάρα πολλοί άλλοι που εμπλέκονται στη στρατηγική. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε και σε μία νέα πρωτοβουλία στα clouds έτσι ώστε ε, να επανέλθει αυτή η στρατηγική για τα clouds. Ίσως αυτά να μην είναι σημαντικά για τις ε, μεταφορές, αλλά αν δείτε λιγάκι την πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών, όλο αυτό το θέμα με το clouding, την ασφάλεια, την προστασία των δεδομένων, όλο αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία. Και να πω τώρα λίγα λόγια για τις μεταφορές. Γιατί βεβαίω και εδώ είμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών, κύριε Πρόεδρε, και αυτή η Επιτροπή έχει μακρά παράδοση στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων. Πολύ μεγάλη σημασία της επιτροπή για την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Να πω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή έχει βοηθήσει ε, στα ERTMS, ε, στον τομέα των μεταφορών. Οι μεταφορές σε μεγάλο βαθμό είναι ένα κομμάτι της ε, ψηφιακής επανάστασης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε χρήση των νέων εξελίξεων στην ψηφιοποίηση. Αν είχα περισσότερο χρόνο, με μεγάλη μου χαρά να σας παρουσιάσω όλα αυτά που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Αλλά βλέπω ότι ο Πρόεδρος με στραβοκοιτάει. Και τώρα να πω κάτι. Όσον αφορά ε, τη χρονική στιγμή που γίνεται η συζήτηση, θέλω να ευχαριστήσω ε, την εισηγήτρια και επίσης ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια που κάνατε. Πάντως μετά από δύο ημέρες... Ε, στο πλαίσιο του, του κινήτου στη Φραγκφούρτη θα υπάρξει και μία ε, συνάντηση των Υπουργών Μεταφορών, το G7, ακριβώς για να εξετάσουν αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι για πρώτη φορά οι Υπουργοί Μεταφορών ε, θα εξετάσουν τις ε, ψηφιακές μεταφορές. Να σας πω, διπλάσιο χρόνο μιλήσατε. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος η συγγήτρια έχει το λόγο. to Κύριε που Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Είναι προφανές ότι έχουμε ενώπιόν μας νέα μοντέλα, νέων υπηρεσιών. Το πρόβλημα ε, δεν είναι η ανάδειξη των νέων αυτών υπηρεσιών, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στα νέα μοντέλα που θα δημιουργηθούν και στις νέες υπηρεσίες. Αν δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο, τότε θα είναι ισότιμο το πεδίο και για όλες τις επιχειρήσεις και η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι ίδια για όλους. Αυτή είναι η πρόκληση που μας περιμένει πρέπει να δημιουργηθεί το απαραίτητο πλαίσιο ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να έχει τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού με όλες οι υπόλοιπες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για το σύντομο των τελικών σας τοποθετήσεων. Ε, λήξη συνεδρίασης 22 Σεπτεμβρίου στις 12 λίγη και η προθεσμία για τις τροπολογίες. Λοιπόν, τελειώνει εδώ η συνεδρία της Επιτροπής πρωινή.